αντί για αντιπρόεδρος θα είμαι πρόεδρος μέχρι τις 4 και 4 περίπου. Ξεκινάμε αμέσως τις εργασίες μας. Ελπίζουμε να έχουμε κόσμο. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να την έχετε μπροστά σας. Έχετε να κάνετε παρατηρήσεις ε, ή διαφωνείτε κάπου. Όχι, άρα θεωρούμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Μία ανακοίνωση. Θα το θυμάστε οι παλιοί, αλλά για τους ε, καινούριου. Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, είχε οργανώσει ένα εργαστήριο υπό την αιγίδα της Αλέν ε, Μακάρθη, της προηγούμενης Προέδρου, για την ε, ασφάλεια των υπηρεσιών συγκεκριμένα στα ξενοδοχεία. Αν Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με αυτό το θέμα, αν και δεν είχε γίνει ποτέ έκθεση. Γι' αυτό ο πρόεδρος, ο κύριος Χάρμπορ, σας ε, προσκαλεί σε ένα γεύμα για την για τα εγκαίνια του εργαστηρίου αύριο υπό την Προεδρία του 12 και 45 με 2 η ώρα το μεσημέρι στο εστιατόριο των μελών, αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο γεύμα είναι προσκεκλημένα. Δεν χρειάζεται να εγγραφεί κανείς έτσι, δεν είναι. Όχι. Καλό θα ήταν να στείλετε ένα email για να γνωρίζουμε πόσο περίσσο άτομα θα είμαστε, για να ενημερώσουμε το εστιατόριο. Περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 8 Φεβρουαρίου. Υπάρχουν αντιρρήσεις, σχόλια. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουν εγκριθεί. Και περνάμε τώρα στη συζήτηση για μια πολύ σημαντική έκθεση ολοκλήρωση της εταιρικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο εισηγητής, ο Αρίας Τσεβερία, είναι φανατικός του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα του δώσουμε λοιπόν το λόγο για όση ώρα χρειάζεται για να παρουσιάσει την έκθεσή του και μετά θα ακούσουμε όλους τους σκιώδεις εισηγητές, κολέγαντε Κάμπος, Κρόσμαν, Τουρούνεν από την ΚΟΕ ποιος είναι σκιώδης. Ο κύριος Γιόγκ. Η κυρία Κλάρκιν και Σαβίνη. Κύριε Τσεβερία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για αυτή την δεύτερη ευκαιρία που προσφέρεται για να παρουσιάσουμε και να δώσουμε τη σημασία στην έκθεση αυτή υποχώνηση που όπως πολύ καλά είπε η Πρόεδρος ε, είναι ε, ευρύτερη. Καθώς ε, ήμουν και συντάκτης ε, για αυτή την έκθεση από πλευρά τη Επιτροπή μα Μελέτησα και εργάστηκα του τελευταίου μήνε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το διασυνοριακό εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή έκθεση είναι το αποτέλεσμα ανάλυση διαφορετικών εγγράφων που αναλύθηκαν για την κατάσταση του εμπορίου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και αρκετών συναντήσεων με του εμπλεκόμενου σε αυτό το τομέα καταναλωτές, επιχειρήσεις ε, και όλους όσους εμπλέκονται στο, στην αγορά online. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς για τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις τους. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κατάφερα να διαπιστώσω ότι είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και είναι διαφορετικά τα προσκόμματα και τα εμπόδια στην ε, ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς online. Οι προκλήσεις στόχοι είναι πολλοί και πολλά πρέπει να γίνουν και είναι απαραίτητα να γίνουν για την ολοκλήρωση της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει το τεράστιο δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει για να βελτιωθούν οι οικονομίες μας. Είναι σημαντικό να εργαστούμε λοιπόν για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό, μια πραγματική αγορά, ευρωπαϊκή αγορά σε αυτό το πεδίο και γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχουμε σαφείς ιδέες και να άγουμε τα προσκόμματα και τα εμπόδια. Και γι' αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα τα πετύχουμε αυτά δημιουργώντας μια κύρια προτεραιότητα για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως τον ηγετικό ρόλο και την πολιτική βούληση για να γίνει αυτό εφικτό, να γίνει δυνατό. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτά τα δύο στοιχεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν επιτέλους η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες από πλευρά στόχων και να το κάνει αυτό με σθένος και ενεργητικότητα. Μπορούμε πολλές εκθέσεις να συντάξουμε και πραγματικά ε, αυτά τα θέματα βρίσκονται επί επί χρόνια. Αλλά δεν θα προχωρήσουμε ποτέ αν δεν έχουμε την πολιτική βούληση να μετατρέψουμε τις ιδέες μας σε πραγματικότητες. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να ξεπεράσει τους σκοπέλους, τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την πρόοδο. Ως Ευρωπαίοι λοιπόν που πιστεύουμε στην ενιαία εσωτερική αγορά πρέπει να έχουμε το αναγκαίο, ας το πω έτσι, φιλόδοξο επίπεδο και να μην πέσουμε στην παγίδα του εθνικισμού και του προστατευτισμού στο οικονομικό πεδίο. Πρέπει να είμαστε ικανοί να καταλήξουμε σε συμφωνίες για να ξεπερνώντας τις μικρές διαφορές, μικροδιαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε ικανοί να υλοποιήσουμε χειροπιαστά τις λύσεις εκείνες που χρειάζεται η Ευρώπη για να ξεπεράσει τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα. Σήμερα <clears throat> είμαστε μπροστά στην εκκίνηση διαφορετικών πρωτοβουλειών που στοχεύουν στο να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Πριν από κάποιες εβδομάδες σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή παρουσιάστηκε η επιπολή διάστημα αναμενόμενη έκθεση του Επιτρόπου Μόντι για τη νέα στρατηγική για την ενιαία εσωτερική αγορά. Στην έκθεση αναγνωρίζεται κυριολεκτικά ότι η ενιαία εσωτερική αγορά online πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της ε, ευρωπαϊκής ψηφιακής ημερήσιας διάταξης για τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια ψηφιακή οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εντόπισε αυτό και το θέσπισε ως μια κυρίαρχη προτεραιότητα και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε υπάρχει ειδικά μονάδα που αφιερώνεται σε αυτό το θέμα υπό την Επίτροπο Κρόης, με την Επίτροπο Κρόης. Και θα έχουμε ευκαιρία αύριο να ανταλλάξουμε απόψεις με την κυρία Κρόης σχετικά. Να βελτιωθεί η κατάσταση διασυνοριακά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρέπει να είναι λοιπόν μια προτεραιότητα για μας. Μια προτεραιότητα που πρέπει με ενεργητικότητα και σθένος να αντιμετωπίσουμε. Όπως εκφράζω και στην έκθεση, στο κείμενό μου, έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να ολοκληρώσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά να βοηθήσουμε την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς. Ένας συντελεστής ε, κύριος μεταξύ αυτών είναι η ανάγκη μιας ενεργούς πολιτικής που θα καθορίζει ότι οι πολίτες, καταναλωτές και επιχειρήσεις θα υποφελούνται πλήρως από την ενιαία εσωτερική αγορά και ότι θα δίνει δυνατότητα αυτό να προσφέρονται προϊόντα και προ, ε, υπηρεσίες καλής αναβαθμισμένης ποιότητας. Πρέπει να δράσουμε λοιπόν για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που θα είναι υποφελές για όλους. Στην σημερινή κατάσταση οικονομικής κρίσης λοιπόν το να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια θα συνεισφέρει χωρίς καμιά αμφιβολία στο να καταπολεμήσουμε την αύξηση των ανισοτήτων και να προστατεύσουμε τους ευάλωτους κανάλτες στα, ε, στους ανθρώπους εκείνους ε, που χρειάζονται υποστήριξη και προστασία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα βοηθήσουμε την οικονομία μας. Η ηλεκτρονική ε, διάσταση του εμπορίου πρέπει να είναι προσπελάσιμη, πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες. Πρέπει να αναζητήσουμε τις πολιτικές που θα καλύψουν τα κενά που υπάρχουν και θα δώσουν την ευκαιρία να δραχθούμε, να δημιουργήσουμε, να εκμεταλλευτούμε το πλήρες δυναμικό στην αγορά online. Πρέπει σε διαφορετικού τομεί να δράσουμε που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και είναι αυτονόητο να ενισχύσουμε πρέπει την εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων που ήδη υφίστανται και ισχύουν. Και όπω ήδη ανέφερα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 17 Μαρτίου και το επανέλαβα σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή στις 28 Απριλίου, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό εμπόριο ισχυρό εσωτερικά που θα μας επιτρέψει να είμαστε και ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι στο εξωτερικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια αγορά online που θα δίνει εμπιστοσύνη από πλευρά των καταναλωτών, που θα διευκολύνει τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και όπου θα προστατεύονται ο ιδιωτικός κόσμος, η ιδιωτική ζωή, τα ε, προσωπικά στοιχεία στις δράσεις μας. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία του 21ου αιώνα αιώνα αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Έχουμε χώρες που διαδραματίζουν έντονα ρόλο και διαγωνίζονται για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο παγκόσμιο. Και έχουμε, παγκόσμια και έχουμε και τις ε, αναδυόμενε τεχνολογίες με επανάσταση χωρίς προηγούμενο και δεν μπορούμε να εξυγχρονίσουμε και να αναθεωρήσουμε την ε, οικονομία μας εκ βάθρων αν δεν προσαρμοστούμε στις νέες αυτές τεχνολογίες ε, και τις προκλήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο και πρέπει να είναι πρότυπο ηγετικό στοιχείο στην παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και να οδηγήσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά στον 21ο αιώνα. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ κάτι για άλλη μια φορά σε μέλη της Επιτροπής, τα έξι σημεία δηλαδή που θεωρώ ότι πρέπει να αναπτυχθούν ή που περισσότερο πρέπει να αναπτυχθούν και πρέπει να εργαστούμε για να βελτιώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο σε αυτά τα σημεία στην Ευρώπη. Και είναι έξι σημεία όπου επικεντρώνεται η προσοχή της έκθεσής μου ακριβώς σε αυτά. Πρώτον, πρέπει να ενισχύσουμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο των χρηστών πανευρωπαϊκά για να μπορούν να αγοράζουν online οι καταναλωτές πρέπει να έχουν ένα αυτοματοποιημένο, μια αυτοματοποιημένη δυνατότητα πρόσβασης. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών στο διαδίκτυο, να βελτιωθεί η ποιότητα, η τιμή και η ταχύτητα του δικτύου όσον αφορά αυτές τις συναλλαγές σε σχέση με άτομα ή χώρες που δεν έχουν την κατάλληλη σύνδεση ακόμα να ξεπεράσουμε την, τον κατακαιρματισμό της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Μεταξύ άλλων είναι αναγκαίο να ενισχύσουμε την εφαρμογή του άρθρου 20 εδαφίου 2 της Οδηγίας περί που απαγορεύει την αρνητική μεταχείριση των ε, ε, πελατών με βάση την εθνικότητα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Τρίτον, πρέπει να ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμένο τρόπο των διατάξεων και ρυθμίσεων. Αυτό θα σημαίνει χωρίς αμφιβολία ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Όχι μόνο όταν θα έρθει η ώρα να συναυθούν συμβάσεις, αλλά και για την επίλυση προβλημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να αναφύονται μεταξύ αγοραστή και πολιτή στι συναλλαγέ. Τέταρτον, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτέ όταν αγοράζουν online ηλεκτρονικά. Πρέπει να καταφέρουμε, πιστεύω εγώ, να κάνουμε συγκεκριμένε δράσει. Πρώτον, την εφαρμογή και υλοποίηση ενό σήματο συμβόλου ποιότητα, ευρωπαϊκού συμβόλου. Επιτήρηση στο διαδίκτυο, εποπτεία και ολοκλήρωση εκστρατιών ενημέρωση, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτε για τα δικαιώματά του. Τα στοιχεία που έχει ένα διαδικτυακό ένας διαδικτυακός τόπος για να μπορεί να έχει εμπιστοσύνη ο καταναλωτής σε αυτές τις συναλλαγές. Ε, ασφαλείς μορφέ ε, πληρωμών κτλ. Επίσης, διασφάλιση της πτυχής της ασφάλειας και των προσωπικών δεδομένων. Πέμπτο, είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες για να δώσουμε κίνητρα στους επιχειρηματίες να εμπορευματοποιούν τα, τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο. Μεταξύ αυτών των πρωτοβουλειών να απλουστεύσουμε τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης όσον αφορά το ΦΠΑ, όσον αφορά τις αγορές, ε, τηλεαγορές, να βελτιωθούν οι μηχανισμοί αγοράς ε, online, να παρουσιάσουμε προτάσεις και λύσεις ε, πρακτικές και εφικτές όσον αφορά και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνουν σε διαφορετικές χώρες ε, οι καταναλωτές. Να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς επίλυσης προβλημάτων μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Έκτο, είναι αναγκαίο να υλοποιήσουμε προσπάθειες που θα γίνουν για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανηλίκων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Πρέπει να εκπονήσουμε τις διατάξεις και ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν ένα υψηλό αναβαθμισμένο επίπεδο προστασίας των ανηλίκων και να έχουμε και την εκστρατεία, εκστρατείες που θα γίνουν για την εξοικείωση και ε, κατάρτιση που θα αφορούν τους γονείς, τους καθηγητές ε, και τους κηδεμόνες με στόχο να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες που έχουν όσον αφορά την εκπαίδευση, την παιδεία, την ε, εκπαίδευση των παιδιών και την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και την αναγκαιότητα να υπάρχει η επιτήρηση, η εποπτεία σε σχέση με τη χρήση του διαδικτύου από παιδιά. Δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω χωρίς να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω πραγματικά την προθυμότητα που υπήρχε από τους χειώδεις εισηγητές για συνεργασία. Με όλες τις προτάσεις και παρεμβάσεις που είχαν και έγιναν την διάρκεια των τελευταίων μηνών, Ήμουν πάντα πρόθυμος να ακούσω τις προτάσεις σας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, που τους ευχαριστώ για τις προτάσεις τους επίσης και τα σχόλιά τους. Και είμαι βέβαιος ότι όλες αυτές σίγουρα θα βρουν την ανταπόκριση την απήχησή τους ε, στη συζήτηση και στην τελική διαμόρφωση αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μας δώσατε τα βασικά σας σημεία, τα εξι 7 σημεία και νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με ποικιλομορφία και αυτό θα βοηθήσει και την έκθεση για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά με σεβασμό και στην ποιότητα των προϊόντων και τις καλές συνθήκες ε, για τις επιχειρήσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε προϊόντα που πουλούνται ηλεκτρονικά τα οποία δεν προσφέρουν ασφάλεια ούτε για τους παραγωγούς ούτε για τους ε, καταναλωτές ενώ επίσης υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα παραποίησης. Ξεκινάμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Campos, παρακαλώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω <clears throat> συγχαίροντας τον συνάδελφο Παύλο Άριας για την παρουσίασή του εδώ και για τις προηγούμενες εισηγήσει ε, για αυτό το θέμα. Είναι ένα κείμενο το οποίο υποβάλλει, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Υπογραμμίζει τα μεγάλα πλεονεκτήματα και όσον αφορά και τις προκλήσεις και τα θέματα που τίθενται για το ηλεκτρονικό εμπόριο για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε καμιά διαφορά ε, σε βάθος στις απόψεις μας και θέλω επίσης να ευχαριστήσω για το ανοιχτό πνεύμα που έδειξε και απέδειξε για να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των stakeholders. Και έτσι <clears throat> μία ε, τέτοια συνάντηση για ενημερωτική που συνέβη και όπου όλοι αποκομίσαμε ωφέλη από αυτές τις επαφές. Θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση θίγει και καλύπτει τα κυριότερα προβλήματα του ηλεκτρονικού ε, εμπορίου. Το θέμα του ΦΠΑ κυρίως, που το στο σκεπτικό και στο σημείο 6 και τα, α, τις δαπάνες που αφορά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς επίσης και θα έπρεπε ίσως κάποια θέματα να τα αναπτύξουμε λίγο περισσότερο. Βλέπουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο ως ένα μέσο για την ικανοποίηση των αναγκών που υπάρχουν για 500 εκατομμύρια καταναλωτές online. Θα θέλαμε όμως οι 500 εκατομμύρια καταναλωτές ε, να είναι διαχειριστές ε, ενός σημαντικού τμήματος του πλούτου στην Ευρώπη. Ένα σημαντικό όπλο για να αναπτυχθεί η ενιαία εσωτερική αγορά μέσα σε μια περίοδο κρίσης οικονομικής. Θα παρουσιάσω τις ε, σκέψεις μου με τη σειρά όπως ε, εμφαίνονται οι παρατηρήσεις της έκθεσης για αυτή την πρόταση. Στο σημείο 4 υπάρχει μια αναφορά σε σχέση με την Επίτροπο Ρέντινγκ, την πρόταση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ε, ροή των πληροφοριών για την σύναψη συμβάσεων. Εδώ υπάρχει μια ιδέα η οποία είναι να έχουμε το μέγιστο εναρμονισμό μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου. Όμως, εγώ πιστεύω σχετικά ότι δεν ξέρω αν πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία ε, σε σχέση με την Επιτροπή. Όπως όταν υπευλήθη ήταν μια πρόθεση από πλευράς Επιτρόπου. Δεν ξέρω αν έχει αυτό το επίσημο καθεστώς για να εμφαίνεται εδώ με την, μετά την ε, ε, διέλευση αυτού του χρόνου. Στο επόμενο σημείο έχουμε την αντιμετώπιση των κανόνων που αφορούν το εμπόριο και τις ε, συμβάσεις online και τις τουριστικές συναλλαγές. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση, όμως συμβαίνει αυτό ακριβώς να είναι το τμήμα του e-commerce, του ηλεκτρονικού εμπορίου, που έχει το περισσότερο αυξηθεί, στο μεγαλύτερο βαθμό αυξηθεί. Και εδώ τι κάνουμε, θα πετάξουμε το μωρό με τα απόνερα του λουτρού, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην υπερρυθμίσουμε ένα τομέα, ακριβώς σε ένα τομέα ο οποίος αυξήθηκε περισσότερο χωρίς κάποιες ρυθμίσεις. Στο σημείο 19 στη συνέχεια, οι υπηρεσίες, ε, ανεξάρτητες υπηρεσίες προστασίας των καταναλωτών είναι μια ιδέα σίγουρα χρήσιμη. Όμως δεν είναι απόλυτα σαφές σε τι στοχεύει. Δεν είναι, εγώ πιστεύω, από τη δική μου ανάγνωση σαφές αν αυτή η ιδέα συγκρούεται με το Solvit ή με κάποιο άλλο μέσο. Έχουμε το Solvit και όλοι έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο Solvit. Ίσως και όλες περισσότερες ελπίδες σε σχέση με τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν. Αν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε ένα νέο θεσμικό όργανο, πρέπει να δικαιολογήσουμε πολύ καλά γιατί θέλουμε να το δημιουργήσουμε. Και η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ίσως θα έπρεπε περισσότερο να ενισχύσουμε αυτά που υπάρχουν σήμερα, για παράδειγμα το Solvit. Φυσικά σε σχέση με το 20 για τις εναλλακτικές δυνατότητες ε, επίλυσης ε, και που πρέπει να ενθαρρυνθούν. Επίσης θεωρούμε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ε, ιδέα το σύμβολο, η σφραγίδα, το σύμβολο ευρωπαϊκής ποιότητας. Και από πλευρά των stakeholders είδαμε την πρόθεση ότι υπάρχουν ομάδες καταναλωτών που δίνουν εμπιστοσύνη σε, για παράδειγμα, ομάδες πολιτών όπου η, η προέλευσή τους, η έδρα τους, η παραγωγή των προϊόντων τους δίνει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές. Αυτή η ιδέα λοιπόν της φραγίδας του, του συμβόλου ευρωπαϊκής ποιότητας είναι ακριβώς μια καλή ιδέα γιατί δίνει τη δυνατότητα αύξησης αυτής της εμπιστοσύνης με την προστασία ακριβώς της ποιότητας. Η ανάγκη του να εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τις ε, πληρωμές online που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, μια και δεν γίνονται δεκτές οι κάρτες, οι τραπεζικές κάρτες, πιστοτικές κάρτες από το εξωτερικό κτλ. Πρέπει να το δούμε αυτό θεωρούμε ότι ο κατακαιρματισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα σημερινά προβλήματα μας οδηγούν στο να επικεντρωνόμαστε στην αποτελεσματικότητα ηλεκτρονικού εμπορίου με σαφείς κανόνες όσον αφορά το ΦΠΑ, κανόνες πληρωμών και δίκαια συστήματα ε, τηλεπληρωμών. Και ίσως ε, να υπάρχει μια μικρή διαφωνία με τον εισηγητή, αλλά όσον αφορά την ε, ενίσχυση της δυνατότητας υποστήριξης για την ε, ε, που φαίνεται κάποιες προτάσεις να είναι ακόμα γενικόλογες ή κάπως ε, αφηρημένες. Ε, ο πυρήνας αυτών των ε, σημείων είναι τα θέματα τα οποία έθιξα εγώ όμως προηγούμενα. Έχουμε και έναν μύτο της Αριάννης ε, που είναι σαφέστερος τώρα σε σχέση με την έκθεση των αιτιολογικών σκέψεων και των σημείων που συμπεριλαμβάνει η έκθεση. Παρότι κάποια σημεία δεν ανταποκρίνονται απόλυτα με τις δικές μας προτεραιότητες στην αλληλουχία, στη συνέχεια που, έχει, που έχουν τύχει. Αλλά αυτά είναι ίσονο σημασία θέματα. Συνοψίζοντας και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω, θέλω να επιβεβαιώσω ότι είχα μεγάλη ευχαρίστηση από αυτή τη συνεργασία με τον εισηγητή. Είναι μια από κοινού θα έλεγα έτσι εισήγηση, συμμεριζόμαστε τις απόψεις του εισηγητή και έτσι τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Merci, Antonio. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κρότσμαν για τους φιλελευθέρους. Α, όχι. Ο φίλος μου, ο κύριος Ροσφόρο. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ να συγχωρήσετε τον κύριο Κρότσμαν, ο οποίος καθυστέρησε εξαιτίας υποχρεώσεων, θα έρθει σε λίγο. Συγχαίρει τον ε, κύριο Αρία για την έκθεσή του. και θα σας ζητήσω το λόγο αργότερα για να κάνω τις δικές μου προσωπικές παρατηρήσεις, για να μην μιλήσω τώρα που μιλάνε οι σκιώδεις συζητητές. Ε, yes, and I will ε, speak. Θα μιλήσω δανέζικα. Προετοιμαστείτε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την έκθεση. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά θετικά σημεία στην έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η διαφάνεια και να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για διακανονισμό διαφορών. Και όλα αυτά τα βλέπουμε στο κείμενο. Να σας επιστήσω την προσοχή στην αιτιολογική σκέψη ΔΕΛΤΑ. Ήδη εδώ και πέντε χρόνια ζητάμε την αναθεώρηση της οδηγίας, γιατί η οδηγία του 2000 είναι μια οδηγία που περιμέναμε για καιρό, αλλά η οποία δεν επαρκεί σε αυτά που μας είχατε υποσχεθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, σε αυτά που μας είχαν υποσχεθεί. Γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο διαθέτει μεγάλο δυναμικό πολλές δυνατότητες για τους καταναλωτές. Όμως πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Είπατε ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαδίκτυο. Θα έπρεπε να θεωρείται δικαίωμα του καταναλωτή και επίσης ότι θα πρέπει αυτή η πρόσβαση να είναι ασφαλής. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ορισμένες σημαντικές αναφορές στο κείμενο. Τώρα, όσον αφορά την πλήρη εναρμόνιση όλων των κανόνων, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν καλό αυτό για τους καταναλωτές. Το συζητήσαμε στην οδηγία για τους καταναλωτές και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες και υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε εναρμόνιση κανόνων Οπότε θα εξετάσουμε αυτή την πιθανότητα, αλλά θα σας πρότεινα να είστε επιφυλακτικοί. Για τα ηλεκτρονικά βιβλία και άλλα ψηφιακά προϊόντα όλο και πιο συχνά απολούνται μέσω διαδικτύου και θα έπρεπε λοιπόν να συζητήσουμε αυτές τις περιπτώσεις σε σχέση με την οδηγία για τους καταναλωτές ζητάει ο εισηγητής περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ε, ενημέρωση για τους καταναλωτές προκειμένου να γνωρίζουν ακριβώς τι αγοράζουν. Επίσης, ζητάτε μια δυνατότητα προσφυγής. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο καλύπτεται και από την οδηγία των καταναλωτών. Και είναι αλήθεια ότι και αυτό το θέμα, εφόσον έχει να κάνει με τους καταναλωτές, πρέπει να το παρακολουθήσουμε στενά. Πρέπει να υπάρξει συνάφεια μεταξύ των δύο κειμένων και σίγουρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο θέμα. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις δικές σας νέες προτάσεις και βεβαίως θα κάνουμε και εμείς κάποιες προτάσεις εκ μέρους της ομάδας μας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντιγιόγκ από την ΚΟΕ. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της ε, δικής μου της ε, πολιτικής ομάδας διότι δυστυχώς ε, χάσαμε τις ε, συζητήσεις ε, που έλαβαν χώρα καθότι ο δικός μας ο δυσηγητής ορίστηκε μόλις τελευταία στιγμή. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να αποφανθεί κανείς επί του θέματος αλλά πράγματι αυτό είναι ένα θέμα όπου πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε και νομίζω αυτό το είπε με απόλυτη σαφήνεια ο εισηγητής. Είναι μια όλο και διευρυνόμενη αγορά. Οι καταναλωτές ε, προσδοκούν, προσβλέπουν σε αυτήν την αγορά. Πρέπει λοιπόν να καταθέσουμε προτάσεις βελτίωσης. Η Κομισιόν πέρυσι ε, προέβησε μια ανακοίνωση και αυτό αναφέρεται στο κείμενο. Γενικά όμως ε, θεωρώ ότι δεν διεκδικούμε αρκετά πράγματα από την Κομισιόν. Δεν θίγουμε το θέμα του χρόνου. Σε ορισμένα άλλα πράγματα εμφανίζεται η στέρηση. Πράγματι υπάρχει κάποια πρόοδος, η κυρία Κρούς έκανε κάποιες προτάσεις για την ε, ψηφιακή ατζέντα, αλλά ε, δεν ε, αρκούν όλα αυτά. Εδώ πρόκειται για εμπορικά συμφέροντα και ως ε, εκ τούτου και λόγω της οικονομικής κρίσης τα συμφέροντα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι ένα γενικότερο μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψουμε προς την κατεύθυνση της Κομισιόν. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα πράγματα θα επιληθούν από μόνα τους. Πάμε σε συγκεκριμένα θέματα, στο copyright. Εδώ πρόκειται για ένα κατακαιρματισμένο σύστημα στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί που εργάζονται και θέλουν να πουλήσουν μουσικά κομμάτια online. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξηγήσουμε, να το αναλύσουμε. Το ίδιο ισχύει και για άλλες μορφές κατάτμησης. Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να εμποδίσουν να πολλούνται προϊόντα ε, διαδικτυακά. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένα καταστήματα που πολλούν αυτά τα προϊόντα. Αυτό ε, εντάξει για τα πολυτελή προϊόντα το καταλαβαίνουμε, αλλά σε άλλα όχι, γιατί αρνούνται τις διαδικτυακές πωλήσει απλά και μόνο για να αυξήσουν τις τιμές. Έτσι λοιπόν πρέπει να καλέσουμε την Κομισιόν να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ λοιπόν θα ήθελα με αυτή την έκθεση να προβάλλουμε περισσότερες διεκδικήσεις. Και θα ήθελα να κάνω και συγκεκριμένες προτάσεις επ' αυτών. Όσο αφορά τώρα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διαδίκτυο. Εδώ πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλη εμπιστοσύνη αυτή από αυτήν που δείχνουν οι καταναλωτέ στα καταστήματα ή η εμπιστοσυνη τους δεν σταματάει στα σύνορα. Πέρα λοιπόν από τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για την προστασία της δικής μας της κοινή αγοράς Ίσως πρέπει να συζητήσουμε και με χώρες όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Γιατί η κατανάλωση αυξάνεται ταχύτατα και ο καταναλωτής ε, δεν ενδιαφέρεται για το κατά πόσο μια χώρα βρίσκεται κοντά ή μακριά. Ε, ο καταναλωτής ε, δεν γνωρίζει πολλές φορές αν μια χώρα δεν είναι αξιόπιστη. Αν παραμείνουμε βέβαια μέσα στην Ευρώπη τότε θα προκαλέσουμε και προστατευτισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς οι ίδιοι επιθυμούμε εξαγωγές σε άλλα μέρη του κόσμου όπου επιθυμούν να αγοράζουν προϊόντα οι καταναλωτές. Αυτή την κατεύθυνση θα θέλαμε να ακολουθήσει η έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you, Madam. Um, and thank you to Mr. Arias for his report. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Αρέας για την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς να συμπεριλάβουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαδικτυακές αγορές. Πρέπει να επωφεληθούμε όλων των ευκαιριών που μας προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο για τους καταναλωτές, όμως επίσης πρέπει να επιτρέψουμε και την ύπαρξη ευελιξία σε αυτή την αγορά για να μην διώξουμε τους καταναλωτές Πρέπει να μειώσουμε τα εμπόδια και για εμένα το πιο σημαντικό είναι η προσβασιμότητα, η δυνατότητα σύνδεσης ε, στο διαδίκτυο προκειμένου να έχουμε κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις και απλό διαδίκτυο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας το τι χρειάζεται ο καταναλωτής. Βεβαίως πρέπει να ανοίξουμε την αγορά σε όλες τις δυνατότητες και να λάβουμε υπόψη μας και τις ανάγκες των πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μαζί με τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Όσον αφορά την αρμόνιση του ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έχω καταστήσει σαφές ότι έχω πολλές επιφυλάξεις και πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω δεν βλέπω επίσης την ανάγκη για μια ανεξάρτητη υπηρεσία. Αυτοί που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο προσπαθούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα τους αρέσει αν πάνε τα χρήματά τους για μια ακόμη υπηρεσία. Και αν έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία τότε δεν θα χρειαστεί αυτή η επιπλέον υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ίσως μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, γιατί αν καταλάβα καλά, ο Αντώνιο θεωρεί ότι υπάρχει και το Solvit, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σαλβίνη, αλλά δεν είναι εδώ. Άρα ο κύριος Τρακόφσκι και με συγχωρείτε για την προσφορά μου, με την προφορά μου. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρέπει να πω ότι η δουλειά ήταν ε, πάρα πολύ καλή. Αν ε, σκεφτεί κανείς πόσο σημαντικό είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, πραγματικά πρέπει να συγχαρούμε τον εισηγητή. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη, στους, να προκαλέσουμε την εμπιστοσύνη εκ μέρους των καταναλωτών στην Ευρώπη. Η διαγωνισμοί ε, online και θα ήθελα να περάσω στα αγγλικά για να είμαι πιο σαφής. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει ε, περάσει αρκετός καιρός ε, και εντωμεταξύ, όπως μας λέει και ο εισηγητής, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έπρεπε να έχει εμφανιστεί εδώ και καιρό η δεύτερη οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχει αλλάξει ο κόσμος από το 2002 με δραματικό τρόπο, κυρίως όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αν πραγματικά ψάχνουμε να ε, βρούμε κάποιες, ε, κάποιους διαγωνισμούς, μηδιωτικού διαγωνισμούς. Ε, το 2002 όταν μιλάγαμε για τέτοιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς είχαμε υπόψη μας κάτι το διαφορετικό. Κυρίως όταν πρόκειται για αυτό που είναι σήμερα το σημαντικότερο μέσο ή ένα από τα σημαντικότερα μέσα για να πουλήσει κανείς προϊόντα στο διαδίκτυο και η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και αυτό είναι σαφές ε, κατά πόσον καλύπτει ε, τους ε, δημόσιους διαγωνισμούς ή όχι. Συμφωνώ με την κυρία Ντεκάμπος ότι δεν πρέπει να προβούμε σε υπερβολικές ρυθμίσεις αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα όπως προτείνει και ο εισηγητής κυρίως όταν πρόκειται ε, για την καλύτερη προστασία των ε, καταναλωτών. Το ποιος φέρει την ευθύνη. Σημαντικό αυτό το θέμα. Παραδείγματο χάρη, στην ε, έκθεση ε, μας λέει ο εισηγητής ότι θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές στον καταναλωτή κατά πόσον ο πολιτής είναι ενδιάμεσος ή τελικός κρίκος. Αυτό είναι σημαντικό για τους διαγωνισμούς. Μερικές φορές δεν ξέρουμε με ποιον ε, έτσι θεωρώ ότι αυτά τα δύο θέματα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω στην έκθεση. Εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες γιατί εκπέμπουμε ένα σημαντικό μήνυμα ότι θέλουμε την επικαιροποίηση αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου και την πραγματικότητα κυρίως στους τομείς που αναφέρθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θα μιλήσουν οι εξή. Κριστέλ και κάποιος από τους τέσσερις μήπως ε, έχει αντίρρηση να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του σκιώδη ηγετή της Άλτε, τον κύριο Κρότσμαν, ο οποίος μόλις έφτασε. Δεν βλέπω κάποιον να διαφωνεί. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια έκθεση η οποία προσπαθεί αυτά που μπορούμε να επιτύχουμε να τα επιτύχει. Και έλαβε χώρα και μια συνάντηση για να ενημερωθούμε για την εμπειρία που έχει προκύψει από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και θέλαμε όλα αυτά να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεση του κυρίου Τσεβερία. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά, θεωρώ ότι εδώ εμείς έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σημαντική ψηφίδα που θα βάλουμε σε αυτό το μοσαϊκό του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες και κυρίως για τις μικρότερες χώρες προσφέρει την ευκαιρία κυρίως στον καταναλωτή να αποκτήσει εμπορεύματα τα οποία δεν παράγονται στην χώρα του. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα ο καταναλωτής να αποκτήσει αυτά τα εμπορεύματα. Αυτό αποτελεί μεγάλη ευκαιρία γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επιληφθούμε του θέματος. Η έκθεση που έχει κατατεθεί αποτελεί μια πολύ καλή βάση και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση επ' αυτής. Το λόγο έχει ο κύριος Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, και εγώ Επιθυμώ να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο για την έκθεσή του. Ε, σε πάρα πολλά ε, σημεία τοποθετεί σωστά το θέμα των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές δεν γνωρίζει κανείς τι θα συντάξουν οι, έκθεση, συνάδελφοι σε μια έκθεσή τους. Εγώ όμως βλέποντας τη έγραψη τον συγχαίρω τον συνάδελφο. Ο συνάδελφος Δεκάμπος διερωτήθηκε κατά πόσο μπορούμε να δεχθούμε την έκθεση γιατί δεν γνωρίζουμε τις ρυθμίσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οδηγία για τον καταναλωτή, νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο μπορούμε να πούμε τι επιθυμούμε και να σκεφτούμε από κοινού μία θέση όπου ε, θέλουμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Αλφιντε Κάμπος. Ε, θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν μπορούσαμε να συζητήσουμε τη συζήτηση με τον συνάδελφο Αρίας ε, το που θέλουμε να καταλήξει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό ισχύει και για την αιτιολογική σκέψη παριθμών 5. Εγώ διαπίστωσα με μεγάλη μου χαρά ότι υπάρχει και μεγάλη προθυμία κυρίως εκεί όπου αναφέρεται ότι ε, θέλει να διευκολύνει τις άμεσες πωλήσει να υπάρχουν οι απαραίτητες εγγύησεις ή ε, ευθύνη για τα προϊόντα και αυτό πέρα από τα σύνορα. Δεν αναφέρεται το πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι ο συνάλφος κύριος Αρίας ε, είναι υπέρ του να δημιουργηθούν οι δυνατότητες να υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο το οποίο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι. Εάν λοιπόν τελικά καταλήξουμε σε κοινή θέση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει και αυτό να επέμβει στην οδηγία για τα δικαιώματα του ε, καταναλωτή. Είναι σαφές ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει ανεξάντλητες ε, δυνατότητες. Εγώ όμως είδα λιγάκι προσεκτικά και την αιτιολογική σκέψη παριθμών 14. Και εκεί καταλήγω στο ότι την επιθυμία του συναδέλφου Αρίας ε, η οποία ε, προφανώς υποστηρίζεται και από τον σκιώδη εισηγητή ε, αυτή την αιτιολογική σκέψη μπορούμε να την εφαρμόσουμε στο βαθμό βέβαια που θα προβλέψουμε και την σχετική πρόβλεψη στην οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Και τώρα θα πω μια μου παρατήρηση. Το υπαριθμόν 17 έχει σχέση με τις online πληρωμές. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί κατ' ουσίαν εδώ έχουμε τρεις βασικές αντιρρήσεις όσον αφορά στις ε, τηλεπολίσεις Πρώτον υπάρχει ε, το, το ο φραγμός ε, της γλώσσας. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εύκολα με οδηγία. Δεύτερον, στις online ε, πληρωμές, παρότι η Ευρώπη θεωρείται ένας ενιαίος χώρος πληρωμών, το πρόβλημα δεν έχει ακόμα λυθεί οριστικά. Και τρίτον, αιτιολογική σκέψη. 17 υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Νομίζω λοιπόν πρέπει να είναι σαφές ότι με ρυθμίσεις αστικής ευθύνης δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το θέμα της απάτης και χωρίς να υπάρχουν ε, ε, κλασικές υποδομές δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Οι υποδομές αυτές θα μεριμνήσουν έτσι ώστε στην ηλεκτρονική αγορά να μην υπάρχουν απάτες προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ε, αγοράς. Και νομίζω ότι εδώ η αστυνομία είναι ο ενδεδειγμένος φορέας για να επέμβει. Άρα δηλαδή πρέπει να αναφέρεται η αστυνομία στην γνωμοδότηση και τελειώνοντας να ευχαριστώ τον συνάδελφο Αρίας. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το κείμενο του κύριου Αρίας είναι πολύ καλό. Είναι σημαντικό που θα ασχοληθούμε, όπως είπε και ο κύριος Σβάμπ, με το θέμα αυτό, τώρα που ασχολούμαστε και με την οδηγία για τους καταναλωτές. Τώρα, ως ε, ευρωβουλευτές οι καινούργοι τώρα κλείνουν ένα χρόνο. Να πω λοιπόν κάτι για τον τίτλο. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε κάποια μέρα να χρησιμοποιήσουμε άλλο όρο και όχι την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η δική μου άποψη είναι ότι ποτέ δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Είναι μια διαδικασία. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε αυτή την ορολογία. Εν πάση περιπτώσει αυτό, ήρθε στο εμπαρόδο το λέω. Τώρα, για εμένα το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πραγματική επανάσταση, γιατί μπορούμε να το δούμε ως επέκταση του κανονικού εμπορίου στις νέες τεχνολογίες, όμως θεωρώ ότι μπαίνουν στην αγορά νέοι φορείς, όχι καταναλωτές, αλλά παραγωγοί οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν ήταν έμποροι. Τώρα γίνονται και έμποροι. Και αυτό είναι που δίνει αυτό το μεγάλο δυναμισμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Γιατί υπάρχει αυτό το κίνητρο να γίνει κάποιος οικονομικός φορέας. Κάτι πολύ σημαντικό προφανώς για όλη την οικονομία μας. Όμως, έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία, έχουμε μεγαλύτερη επιλογή, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να σημαίνει λιγότερα δικαιώματα, ειδικά για τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν διεξάγεται καλώς. Και ειδικά όταν πρόκειται για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό θα έπρεπε να είναι το σημείο εκκίνησής μας. Δύο πράγματα τώρα για συγκεκριμένες παραγράφους. Για την 24. Όσον αφορά τις ετικέτες εμπιστοσύνης. Ήδη το ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι. Αύριο θα αναπτυχθεί περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και όσο περισσότερο αναπτύσσεται, τόσο περισσότερο θα βλέπουμε ιστοσελίδες τόσο εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αραβικών, αμερικανικών κτλ θα ήταν προστατευτισμός, γιατί εγώ δεν νομίζω, να κάνουμε αυτή την εργασία εναρμόνισης και αύξησης της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς. Και αυτή τη δουλειά να την καταστήσουμε ορατή στο σύνολό των καταναλωτών. Να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να έχετε περισσότερη εμπιστοσύνη. Και αυτό θα πρέπει κάπως να το βλέπουν και στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, όλη αυτή η δουλειά που θα κάνουμε για την εσωτερική αγορά θα κινδυνεύει εξαιτίας παραδειγμάτων αρνητικών σε περιπτώσεις ε, εμπορίου εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε και για μια ετικέτα οικολογικής εμπιστοσύνης. Εγώ θα ήθελα και μια ετικέτα εμπιστοσύνης για το ηλεκτρονικό εμπόριο που να δείχνει ότι υπάρχει κάποια δέσμευση από αυτούς τους φορείς. Και δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί προστατευτισμός. Και το δεύτερο σημείο, κοιτάξτε, εγώ βρίσκομαι σε μία χώρα, α, για το σημείο 10, όχι συγγνώμη, δεν θυμάμαι πού. Στη χώρα μου, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε μαγαζί με φυσική υπόσταση για να κάνουμε ηλεκτρονικό εμπόριο. Και είμαι ευνοϊκός στο να μην υπάρχει τέτοιος περιορισμός, όμως θα ήταν ενδιαφέρον να εξετάσουμε την τυπολογία. Και να δούμε ότι υπάρχουν ηλεκτρονικές δραστηριότητες που γίνονται χωρίς φυσική έδρα, αλλά και περιπτώσεις όπου έχουμε συμπληρωματική δράση ηλεκτρονικού εμπορίου και συμβατικών πωλήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να έχει δυνατότητα επιλογής ο καταναλωτής και κάπου θα έπρεπε να φαίνεται αυτό. Τέλος, υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, διάδοση του γρήγορου διαδικτύου Μίλησε ο κύριος Αρίας για μία ανεξάρτητη υπηρεσία. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να έχουμε κάποιο είδους παρακολούθησης ή κάτι άλλο που θα επέτρεπε στους καταναλωτές που δεν γνωρίζουν ακόμη πώς λειτουργεί το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο να συνοδεύονται στα πρώτα τους βήματα σε αυτό με κάποιο είδου εκστρατεία ή κάτι άλλο αντίστοιχο που θα τους ε, επιτρέψει αυτό. Ευχαριστώ Ρομπέρ. Ζητάμε πολλά χρήματα για εκστρατείας πληροφορίας και κατάρτισης. Δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να κάνουμε στο μέλλον. Και όσον αφορά την ευρωπαϊκή ορολογία, ολοκλήρωση της αγοράς κτλ είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί όροι που δεν καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και τους οποίους χρησιμοποιούμε εμείς. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να αλλάξουμε λίγο το λεξιλόγιο. Κριστέλ παρακαλώ. Να κάνω κάποια σύντομα σχόλια για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όλοι μας νομίζω ότι καταναλώνουμε προϊόντα ηλεκτρονικά, άρα μας ενδιαφέρει όλους αυτό το θέμα. Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να επιληθούν στο πλαίσιο της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι σημαντικό όμως οι καταναλωτές να μπορούν να εμπιστεύονται τις αγορές από το διαδίκτυο είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό για τον καταναλωτή από το να υπάρξει εναρμόνιση των κανόνων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι είναι λιγότερο σημαντικό για τους καταναλωτές. Και αυτό φαίνεται σαφώς στο σημείο 17 που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικό. Το βασικό είναι να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη. Άρα, όταν ένας ε, καταναλωτής έχετε στο δικό μας δικαστήριο για να κάνει μια προσφυγή για μια ιστοσελίδα γερμανική, τα πράγματα περιπλέκονται και περνάνε έξι μήνες μέχρι να καταλήξει το δικαστήριο σε απόφαση. Αυτό είναι πολύ. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι βέβαιος για το σεβασμό των κανόνων ο καταναλωτής. Πρέπει λοιπόν να τους προσφέρουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Όσον αφορά το 24 και τις ετικέτες εμπιστοσύνης, στη Δανία έχουμε ένα τέτοιο είδος ετικέτες που επιτρέπει στους καταναλωτές να εμπιστεύονται περισσότερο κάποιες ιστοσελίδες στο ίντερνετ. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η λύση, γιατί επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη. Θα έπρεπε βεβαίως εκεί να εμπλακούν οι δημόσιες αρχές για να πιστοποιούν αυτούς που θα φέρουν την ετικέτα. Ευχαριστώ Κριστέλ. Ένα ερώτημα για τον κύριο Τρασκόφσκι. Σας πειράζει για 10 λεπτά να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν μετά την Εύελιν που έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Στασκόσκη που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Παρότι και το θέμα της Ελβετίας και της ΕΕ είναι σημαντικό σίγουρα και αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν για μια πολύ καλή πρόταση που ο κύριος Άριας μας έκανε εδώ με την έκθεσή του με βάση την οποία πολύ καλά μπορούμε να εργαστούμε και όπως και οι συνάδελφοί μου κάποια σημεία ήθελα να επιλέξω τα οποία τα θεωρώ ιδιαίτερα θετικά. Ήθελα να πω στον κύριο Ροσφό το σημείο 10 στο δεύτερο τμήμα όπου υπάρχει η δέσμευση της, ε, ε, των συναλλαγών online. Νομίζω είναι ένα σωστό αίτημα αυτό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ε, των συναλλαγών και δεν θα έπρεπε να επιβάλλουμε κάτι το οποίο επιτρέπεται και κάτι άλλο το οποίο δεν επιτρέπεται και πρέπει να το αφήσουμε σε ένα ανοιχτό και διαφανές πλαίσιο να γίνονται οι συναλλαγές. Ακριβώς όπως και εμείς δεν θέλουμε να δεσμεύσουμε τους καταναλωτές να κινούνται υποχρεωτικά online όταν θέλουν να αγοράσουν κάτι. Και αν κάποιος πει «Ε, δεν θέλω να αγοράσω μέσω ίντερνετ, μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται να το κάνουν και αυτοί δεν υποχρεώνονται να αγοράζουν online ηλεκτρονικά. Μην το ξεχνάμε λοιπόν ότι πρέπει ο καθένας να αποφασίζει ελεύθερα ο ίδιος τι θα κάνει και πώς θα κινείται. Ήθελα να πω ότι το σημείο 17 μου αρέσει και εμένα ιδιαίτερα. Διότι ως θέμα αρχής αναφέρεται στα προβλήματα εκείνα που πολλοί καταναλωτές αντιμετωπίζουν και που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, με τρόπο ώστε με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό ώστε στην τελική ρύθμιση αν θα έχουμε ε, μια ιδιωτική προσαρμογή όχι δεν είναι αυτό το πρόβλημα το πρόβλημα είναι να δούμε ότι πρέπει τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το δει και ζητούμε αυτό ακριβώς να ε, προαχθεί και να επιληθεί και πρέπει να δούμε ενισχυμένα περισσότερο στο κείμενό σας κύριε Άρια, αυτό το οποίο αναφέρατε, το θέμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μέσω του διαδικτύου πάρα πολλά στοιχεία δίνονται, προσωπικά στοιχεία, είτε πληρώνοντας ο αγοραστής, είτε με άλλο τρόπο. Η προστασία αυτών των προσωπικών δεδομένων και η αυτοδιάθεση από πλευράς των δικαιούχων αυτών των στοιχείων είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να αναφέρω ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε από κάποιον άλλο πιο πριν και που θεωρώ όμως πολύ θετικό και σημαντικό. Είναι το είναι 21 αυτό, όπου πρόκειται για ένα μεγάλο ή μέγιστο βαθμό ασφάλειας για τους ανηλίκους που θέλουμε να διασφαλίσουμε. Στη σημερινή εποχή που όλο και περισσότερες συναλλαγές όχι μόνο μέσω ε, ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και μέσω κινητού τηλεφώνου. Τώρα έχουμε και το iPod και δυνατότητες πολύ ευκολότερης πρόσβασης και για νεότερα άτομα και για ανηλίκους. Να σκεφτούμε υποχρεωτικά λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα προσφέρουμε προστασία για τους ανήλικους, ε, για αυτούς τους νέους ε, που πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία αυτή και τι θα κάνουμε. Ξέρω στη δεκαετία του 80 και στη δεκαετία του 90 είχαμε επίμαχη συζήτηση με έντονο τρόπο στην Γερμανία για τις αγορές στον δρόμο προς ανηλίκους και όπου οι κανόνες δεν τι ετηρούνται όταν, σε σχέση με το ότι δεν έπρεπε να συνάπτουν τέτοιου είδους συναλλαγές σε σχέση με ανηλίκους. Μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το πρόβλημα ακόμα ενισχυμένα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να αναφαίνεται, να, να ξαναφανεί διότι δεν έχει απέναντί του κανείς ε, τον, ε, πολιτι... τον αγοραστή, με συγχωρείτε, ο, ο, όποιος συναλλάσσεται στο διαδίκτυο και δεν ξέρει αν έχει κάποιον ανήλικο μπροστά του ή κάποιον άλλο. Για προστα... προστασία λοιπόν των ε, συναλλαγών αυτών θα πρέπει να υπάρξει κάποιο σύστημα ώστε να μην συνάπτονται τέτοιου είδους συναλλαγές που δεν θα είναι νόμιμες. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό το σημείο 21 πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ευχαριστώ. Πρόκειται για θέμα επί του οποίου πρέπει να εμβαθύνουμε. Ενδιαφέρει και τις επόμενες γενές. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Νταβίτ Μάιερ που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΓΑΜΑ ΣΑΝΚΟ. Πράγματι, εγώ εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ, αλλά θέλω να πω ότι η ε, έκθεσή μας ε, είναι το αποτέλεσμα πολλών υπηρεσιών της ε, Κομισιόν και εμπίπτει στην ευθύνη πολλών ε, τομέων. Θα ήθελα ε, να κάνω τρεις παρατηρήσεις βασικά σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αφορά μόνο αυτό. Δηλαδή, αν το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί και αντιμετωπίζεται ως πραγματική εναλλακτική λύση για τους καταναλωτές, για τις αγορές τους, τότε έχει και πάρα πολλές επιπτώσεις, θετικές προεκτάσεις στο λιανικό εμπόριο, το οποίο και μπορεί να βελτιώσει. Ήδη γνωρίζουμε ότι ε, τα καταστήματα offline, τα φυσικά μαγαζιά, εξετάζουν το τι προσφέρεται διαδικτυακά. Διότι οι ε, καταναλωτές ψάχνουν όλο και περισσότερο το τι υπάρχει διαδικτυακά. Μετά πάνε σε ένα μαγαζί ε, και ρωτάνε πόσο κάνει αυτό, μπορώ να το βρω στην τάδε τιμή στο διαδίκτυο. Αυτό μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αγοράζουν ε, πράγματα διαδικτυακά. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να γίνει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Και τότε υπάρχουν πάρα πολλά πλονεκτήματα. Καλύτερος ανταγωνισμός, καλύτερη λειτουργία της αγοράς που ε, έχει θετικές, όπως σας είπα, προεκτάσεις και στα φυσικά μαγαζιά. Ο καταναλωτής θα αποφεληθεί τα μάλα εάν τελικά βελτιώσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Διότι οι αγορές για τα ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες ε, θα γίνουν πιο ολοκληρωμένες. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν πρέπει να θεωρείτε ότι είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό ε, παράλληλο με την οικονομία μας, γιατί ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται τα καταστήματα και οι καταναλωτές ε, κατά κάποιον ε, τρόπο αποστασιοποιούνται γιατί προκύπτουν πάρα πολλά ωφέλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ηλεκτρονικό εμπόριο να λειτουργεί διασυνοριακά και αυτή είναι η πεμπτουσία της έκθεσης της Κομισιόν γιατί βλέπουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, αυξάνεται σε σταθερό ρυθμό, όμως το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν επεκτείνεται. Δεν λειτουργεί αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι οι επιχειρήσεις αρνούνται να πουλήσουν διασυνοριακά στους καταναλωτές. Εάν λοιπόν λειτουργούσε το διασυνοριακό εμπόριο, τότε τα θετικά αυτά αποτελέσματα από το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορούσαν να επεκταθούν στο σύνολο της ε, κοινή ε, αγοράς. Αντί δηλαδή να έχουμε υψηλές τιμές στο λιανικό εμπόριο σε ορισμένα κρατημέλη και περιορισμένη προσφορά, Εάν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο καταστεί μια αξιόπιστη λύση για ένα καταναλωτή σε μια συγκεκριμένη χώρα, τότε καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει να αγοράζει διαδικτυακά και τότε το λιανικό εμπόριο της χώρας του θα πρέπει να προσαρμοστεί, να βελτιώσει την προσφορά του. Γι' αυτό λοιπόν το να λειτουργήσει το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι καθοριστική σημασία, όχι γιατί θέλουμε οι καταναλωτές όλο και περισσότερο να αγοράζουν διαδικτυακά, αλλά γιατί σας λέω θα έχει πολύ θετικές επιπτώσεις στο σύνολο του λιανικού εμπορίου, κυρίως στα μικρότερα και τα μεσαίου μεγέθους κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν τα μεγάλα κράτη-μέλη όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αρκετά επεκταμένο, σε άλλα πάλι όχι. Ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπο να ολοκληρώσουμε την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα επωφελές και για τους ε, καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στα κράτη-μέλη. Το τρίτο που θέλω να πω είναι το εξής. Η έκθεση της Επιτροπής λέει ότι το γιατί δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο αυτό είναι ένα περίπλοκο θέμα και υπάρχουν πάρα πολλά που εμποδίζουν τι εταιρείε να προσφέρουν διασυνοριακά. Νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι σε σχέση με πριν από 5 ή 10 χρόνια, τώρα το πρόβλημα δεν είναι τόσο η αξιοπιστία του καταναλωτή, η οποία ε, ενισχύεται όλο και περισσότερο. Το πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα στη διασυνοριακή αγορά είναι ότι οι εταιρείε αρνούνται να απολύσουν. Έχουμε περίπου κάνει 13.500 συναλλαγές και στα 27 κράτη-μέλη και ε, πάνω από το 61% των περιπτώσεων, σε πάνω από 61% αρνήθηκαν οι εταιρείε να πουλήσουν. Εάν λοιπόν δεν ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, τότε το θέμα ε, τη εμπιστοσύνη του καταναλωτή και λέω δεν υφίσταται. Αφού δεν υπάρχει τίποτα να αγοράσει, ποιο να εμπιστεύεται. Ω εκ τούτου, αυτά τα θέματα πρέπει να ερευνήσουμε. Γιατί δηλαδή αρνούνται οι εταιρείε να πουλήσουν διασυνοριακά. Βεβαίω και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. βεβαίω και υψηλή ε, προστασία, αλλά εναρμόνιση για να είμαστε σίγουροι ότι οι εταιρείε είναι πρόθυμες να πουλήσουν το θέμα της προστασίας, αυτό είναι που βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις πίσω από το 61%. Ε, και βεβαίως ε, θέλουν οι καταναλωτές αποτελεσματική ενημέρωση, προστασία και κυρίως ε, μηχανισμούς αποζημίωσης. Αν δηλαδή τα πράγματα δεν πάνε καλά, να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι θα βρεθεί μια εύκολη λύση να αποζημιωθούν. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε και να ακούσουμε τα συμπεράσματα από αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση, θα ακούσουμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που μίλησαν σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και για τα σχόλια τους, τα καλά τους σχόλια για την έκθεσή μου. Ακούσαμε πολλές υποδείξεις, προφορικές τροπολογίες αν θέλετε, για διάφορα σημεία του εγγράφου. Νομίζω όμως ότι πολλά από αυτά τα θέματα ήδη καλύπτονται από το έγγραφο. Το έγγραφο βεβαίως είναι εξ ανάγκης σύντομο, αν και παραμένει ανοιχτό σε τροπολογίες. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι αρκετά ανοιχτό. Εν πάση περιπτώσει, πολλές από τις τροπολογίες είναι ευπρόσθεκτες. Θα ήθελα εδώ πάντως να τονίσω ότι όπως είπαν και άλλοι, το πολύ σημαντικό θέμα είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και για να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης πρέπει να προσφέρουμε πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τις συναλλαγές που πρόκειται να διεξάγουν, ειδικά αν πρόκειται για διασυνοριακές συναλλαγές. Είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι πληρώνουν, πώς το πληρώνουν, τι αγοράζουν να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται για πειρατικό ή παραποιημένο προϊόν και ότι καλύπτεται από όλες τις εγγυήσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλά και η Εθνική βεβαίως. Ένας άλλος τρόπος να αυξηθεί η εμπιστοσύνη είναι με αύξηση της ασφάλειας πληρωμών. Και η παροχή δυνατότητας για την επίλυση διαφορών. Επίσης, όπως είπα και πριν, πρέπει να είναι σίγουροι οι καταναλωτές ότι πληρώνουν νόμιμα προϊόντα. Τώρα, το αν χρειαζόμαστε ειδική εκπαίδευση δεν ξέρω. Είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγα χρόνια η βασική σχολική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες. Ήδη γίνεται αυτό σε κάποιες χώρες και υποθέτω ότι στα μαθήματα πληροφορικής θα γίνεται λόγος και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό που όμως πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μάθουμε τους καταναλωτές να φέρουμε πιο κοντά σε αυτούς το ηλεκτρονικό εμπόριο, να συνειδητοποιήσουν ότι είναι κάτι το απλό, κάτι το καλό για αυτούς. Και συμπερασματικά, δεν νομίζω ότι η δική μας γενιά θα είναι η γενιά που θα χρησιμοποιήσει τόσο πολύ τις ηλεκτρονικές αγορές. Η γενιά των παιδιών μας όμως θα χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο για τα ψώνια της και τις αγορές της. Τα παιδιά μας που είναι παιδιά σήμερα, όταν ενηλικιωθούν θα ζουν σε έναν κόσμο όπου καθημερινά θα κάνουν τέτοιου είδους συναλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άριας. Είχαμε μια επικοδομητική συζήτηση και υποθέτω ότι θα υπάρξουν και τροπολογίες. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 8 Ιουνίου 16 το απόγευμα, 4 το απόγευμα. Κύριε Αρίας, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ε, το Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, επιτρέψτε μόνο αυτό να πω, για το χρόνο που βρήκε για μας. Για να μην χάνουμε χρόνο, δεν επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες. Περνάμε σε μία δεύτερη έκθεση εξίσου σημαντική και εδώ θα χαρεί ο κύριος Ροσφόρ γιατί δεν μιλάμε για ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά για accomplishment, για επιτυχία. Έχει το λόγο ο εισηγητής ο κύριος Τρασκόφσκι για να μας μιλήσει για τους στόχους του. Και μας συγχωρείτε που σας καθυστερήσαμε. Είναι η τρίτη φορά που το συζητάμε το θέμα, όχι η πρώτη, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, ε, θα μιλήσουμε για την εσωτερική αγορά στην Ελβετία και νομίζω αυτό το θέμα αποφασίσαμε θα μιλήσουμε κυρίως για τα εμπόδια που υπάρχουν στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ε, ε, την, ε, στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετίας. Ε, να πω λοιπόν το εξή πρώτα απ' όλα. Μιλήσαμε σχεδόν με όλους, ε, μιλήσαμε με τους βουλευτές στη Βέρνη, μιλήσαμε με τον ε, πρόεδρο του καντονίου της Βέρνης. Μιλήσαμε επίσης και με τον πρόεδρο της χώρας για να καταλάβουμε λιγάκι την ελβετική άποψη. Και κατ' ουσίαν όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε, δουλεύουμε πάνω στο θέμα αυτό τους τελευταίους μήνες. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, έχουν προκύψει δύο διαφορετικές ε, προσεγγίσεις, γιατί είχαμε πάρα πολλές διαβουλεύσεις. Είχαμε διαβουλεύσεις με επιτροπές, με επιχειρηματίες και πολλούς άλλους. Και όταν μιλάει κανείς με τους Ελβετούς ε, συναδέλφους, πολλές φορές την κανείς να πιστέψει ότι είναι περιττή η κουβέντα, γιατί πολλοί από τους συνομιλητές μας λένε ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με την κατάσταση και δεν περιμένουν τίποτα το σπουδαίο. Βεβαίως, ε, και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές ακούμε να μας λένε ότι θα πρέπει καλύτερα να ε, επιδιώξουμε μια τελείως διαφορετική σχέση και να προσεγγίσουμε τους ελευθερούς συναδέλφους με μία προσέγγιση της τάξης ε, είτε αν, αν σας αρέσει καλός, αν δεν σας αρέσει κακός. Πάντως ε, τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε στις σχέσεις μας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας απορρέουν από το ότι οι σχέσεις είναι πολύ περίπλοκες και αυτό απορρέει και πάλι από το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μυστήρια και περίεργη συμφωνία. Η Ελβετοί ήταν εκείνοι που διαπραγματεύτηκαν, επιθυμούσαν διακάως αυτή την ε, συμφωνία, κατά κάποιον τρόπο την εφήβραν και όλες, μετά όμως την απέρριψαν οι πολίτες αυτή τη συμφωνία των ελβετικών αρχών. Και τελικά καταλήξαμε σε μια ρεαλιστική ε, λύση. Δηλαδή είδαμε το καθεστώς και σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί τρόποι για το πώς μπορεί να βελτιώσει μια κατάσταση. Και θα σας πω λίγα πράγματα γιατί τα περισσότερα βρίσκονται στην έκθεσή μου. Εξετάσαμε λοιπόν ε, τα μέτρα υποστήριξης ε, που παρουσιάζει η Ελβετία και καταλήξαμε στο ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσουμε τους Ελβετού συναδέλφου, ότι σημαντικότερο είναι τα, να υπάρχει αναλογικότητα. Γιατί αλλιώ δεν υπάρχει νομική ασφάλεια στην αγορά. Όσον αφορά στο θέμα της ε, παρεμπόδιση υλοποίησης της κοινή αγοράς, ε, αυτό το θέμα ε, εμφανίστηκε και στη δική μας την πλευρά και γι' αυτό προτείνουμε να υπάρξει κάποια αναθεώρηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ενιαία εφαρμογή των κανόνων περί κοινή αγοράς. Δύσκολο αυτό σε διμερές επίπεδο, όμως ε, σε αυτό θα πρέπει να προσβλέπουμε. Γιατί αν δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή κανόνων, δεν υπάρχει και νομική ασφάλεια. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία ευελιξίας, κυρίως όσον αφορά ε, στην ταχύ εφαρμογή ρυθμίσεων περί ατόμων. Ε, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς είναι δυνατόν να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός, κυρίως όσον αφορά στην εφαρμογή των αποφάσεων. Μπορούν να υπάρξουν τρόποι ε, για να συμμετέχουν και οι Ελβετοί στη λήψη των αποφάσεων. Μιλώντας βέβαια στους Ελβετούς συναδέλφου, αλλά σκεπτόμενοι και τα δικά μας στην ευρωπαϊκή πλευρά, ακόμα και αν καταλήξουμε στο ότι προς το παρόν τουλάχιστον μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στο status quo και να βελτιώσουμε τις ε, διμερείς σχέσεις, ε, νομίζω ότι θα προκύψουν τεράστια θέματα και οι Ελβετοί συνάδελφοι γνωρίζουν αυτή την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να σας τα παριθμίσω, αλλά είναι το πακέτο για τα εμπορεύματα, τα δικαιώματα του καταναλωτή, ε, δημόσιοι ε, διαγωνισμοί, οτιδήποτε αγγίζει κανείς, ηλεκτρονικό εμπόριο. Εμείς έχουμε πάρα πολλά να θίξουμε και κυρίως αν δει κανείς τις ε, διμερείς σχέσεις μεταξύ ημών και της Ελβετίας, καταλήγει στο ότι είναι σχεδόν αδύνατον να προχωρήσει κανείς στη βελτίωση των σχέσεων χωρίς να αγγίξει αυτά τα καυτά θέματα. Θεωρώ λοιπόν ότι μιλώντας με τους συναδέλφους και έχοντας ακούσει την ε, άποψη της Επιτροπής κατέληξα στο ότι τουλάχιστον όσον αφορά στο μέλλον θα πρέπει να αναζητήσουμε, να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να μπορέσουμε να υπογράψουμε μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να λύσουμε όλα τα θέματα ε, τα οποία θα τοποθετηθούν επιτάπητος ε, στο εγγύς μέλλον. Προφανώς θα πρέπει να ε, πρόκειται για συγκεκριμένες συμφωνίες επιμέρους συμφωνίες, εμείς ε, στο σχέδιο που έχουμε καταρτήσει εξηγούμε ότι πρέπει να διερευνηθούν αυτές οι δυνατότητες. Και νομίζω, <clears throat> όπως σας είπα, ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι να μην πάμε στους Ελβετούς και να τους κάνουμε κήρυγμα, αλλά να ακούμε τι έχουν και αυτοί να μας πούν, να τους δώσουμε την εντύπωση ότι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια ιδιότυπη σχέση, η οποία χρήζει και ιδιαίτερης προσοχής και από τις δύο πλευρές. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι η περίπτωση μιας χώρας που ε, θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια άλλη περίπτωση όπου πρέπει να βρούμε κάποιες προσαρμοσμένε ε, λύσεις. Ε, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει ε, να δείξουμε στους συνομολητές μας ότι υπάρχει και άλλο συνομολητής, το Κοινοβούλιο γιατί υπάρχει βέβαια η Επιτροπή που είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων, όμως είναι απαραίτητο και οι βουλευτές ε, να διεξάγουν διάλογο. Οι Ελβετοί συνάδελφοι εκτιμούν ιδιαίτερα το ότι μια Επιτροπή του Κοινοβουλίου ασχολείται με το δικό τους το θέμα. Η καταληκτική μερομηνία για την υποβολή τροπολογιών πλησιάζει πολύ γρήγορα μετά την ακρόαση και μετά την επίσκεψη και εγώ ίδιος ε, θέλω να αλλάξω την έκθεσή μου, αλλά περιμένω και τις τροπολογίες που ενδεχομένω ε, κατατεθούν. Θα συνεργαστώ με τους σκιώδεις εισηγητές για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ε, συμβαστικές προτάσεις. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία που βοήθησε στο να οργανωθεί η ακρόαση και αυτό το τόσο σημαντικό ταξίδι στην Ελβετία. Βεβαίως ε, και υπήρχαν προηγούμενα, αλλά αυτό αποτελεί ένα ε, ορόσημο για μας ε, για το μέλλον. Ευχαριστώ τους ηγητές και θεωρώ ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορέσουμε τελικά να κλείσουμε το θέμα μέσα από τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Το η πρώτη πρόκληση για την Προεδρία μου ήταν να πω το όνομά μου, αλλά το, το όνομά σας με συγχωρείτε, αλλά το επόμενο όνομα δεν είναι δύσκολο γιατί είναι φιλανδικό, ο κύριος ε, Ρίπον που σημαίνει αλεπού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τρασκόφσκι για την ισορροπημένη του έκθεση. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή διαφωτίζει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΕΟΧ. Ε, Έχαμε κάνει πολλές συνεδριάσεις και πολλές διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η συμφωνία με την Ορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενστάιν είναι η ευκολότερη εναλλακτική λύση οι Ελβετοί αποφάσισαν να μην υπογράψουν τη συμφωνία και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σεβαστούμε. Ακόμη και αν αυτό δεν είναι εύκολο για εμάς. Η σύσταση για διμερείς σχέσεις είναι θετική. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε να προσιλητήσουμε τους Ελβετούς. Απλά πρέπει να δείξουμε κατανόηση στις θέσεις τους. Για το πλαίσιο αυτό καθ' αυτό της ε, συνεδρίασης δεν έχω να πω κάτι επιπλέον. Όμως, να μιλήσω λίγο για τις προκλήσεις αυτής της συμφωνίας. Μια μεγάλη πρόκληση είναι η πολύ αργή εφαρμογή της συμφωνίας για λόγους ε, θεσμικούς και διαρθρωτικούς που έχουν να κάνουν με τη συμφωνία ΕΟΧ. Θα έπρεπε να μειώσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσει η εφαρμογή μιας συμφωνίας από τη στιγμή της έγκρισής της. τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς. Είτε πρόκειται για την οδηγία για τις υπηρεσίες, είτε για άλλες οδηγίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρόιτσμαν και πάλι εκ μέρους της UN. Man, der Bericht äh, Κοιτάξτε, ε, είναι πράγματι δύσκολο με να πετύχει κανεί μερικά πράγματα. Έξι με την ε, Νορβηγία, Λίχτενστάιν, αυτά δεν δημιουργούν προβλήματα. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίω εδώ είναι η σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία. Ο εισηγητή περιορίστηκε ε, σε αυτό και μόνο και νομίζω ότι καλά έκανε. Ε, σημασία έχει τελικά ε, να δείξει κανείς τα προβλήματα που υπάρχουν κυρίως κατά την εφαρμογή της οδηγίας ε, παροχής, περιπαροχής υπηρεσιών. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελβετία. Να περιγραφούν λοιπόν τα προβλήματα, να παρουσιαστούν κάποιες λύσεις. Αυτό είναι αξιέπαινος ο εισηγητής που το έπραξε. Κατά τα άλλα το έδειξαν αυτό και οι ακροάσεις, ε, το έδειξαν και οι συζητήσεις με τους ε, βουλευτές ε, της Ελβετίας. Είδαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελβετία. Γιατί η Ελβετία έχει μια τέτοια δομή που δεν επιτρέπει καν να υιοθετεί η Ελβετία αυτά που εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελβετία θα μπορούσε κανείς να πει ε, να, υιοθετήστε τι οδηγίε, υιοθετήστε τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν γίνεται όμω αυτό γιατί στην Ελβετία δεν υπάρχει ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο όπω υπάρχει α πούμε στη Γερμανία το οποίο να μπορεί να ελέγξει την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Ξέρετε ότι στην Ελβετία ε, με την μορφή δημοκρατία που υπάρχει στη χώρα αυτή ο λαό είναι εκείνο που αποφασίζει τελικά μέσα από τα δημοψηφίσματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να πει κανεί στην Ελβετία, ξέρετε κάτι, υιοθετήστε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και γι' αυτό το αναγνωρίσαμε αυτό και θεωρώ ότι είναι καλό που περιοριζόμαστε σε αυτά που είναι εφικτά για να επιτευχθεί βελτίωση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας. Αυτό εξάλλου αναφέρει και η έκθεση. Εγώ ε, σκέφτηκα πάρα πολύ κατά πόσον θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε περαιτέρω τη σχεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας. Κατέληξα όμως ε, στο συμπέρασμα ότι πέρα από αυτά που προτείνει η έκθεση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όσον αφορά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Και δεν μπορούμε γιατί από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει τελείως διαφορετική δομή από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν τούτου η έκθεση είναι ιδιαίτερα ισόρροπη, Η Ελβετία έκανε και αυτή κάποιες ε, παραχωρήσεις και στην ε, αρχή αναφέρονται ποια είναι τα προβλήματα στην αρχή της έκθεσης. Ε, την έκθεση βρίσκω ιδιαίτερα ισόρροπη και δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες στην έκθεση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το ότι άμβλυνε τους τόνους γιατί αν δεν είχε προβεί σε αυτή την άμβλυνση των ε, προβλημάτων ε, θα επικρατούσε δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο με βάση αυτά που υφίσατε μπορούμε να επιτύχουμε περαιτέρω βελτίωση. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Επόμενος, επόμενη εισηγήτρια ερωτώσα μάλλον, κυρία Μιλλέρ. Θέλω να πω ότι εμείς ε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα, λέει η κυρία Ρούλε. Εμείς ε, είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις με πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες. Φαίνονται όλα αυτά στην έκθεση και δεν υπάρχει κανένα κενό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο πρόεδρός μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που αναλάβατε την Προεδρία γιατί εγώ ήμουν στην αντιπροσωπεία με το Ιαπωνικό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι είναι σημαντικό να κρατήσουμε στενές σχέσεις μαζί τους. Καταρχάς, ε, επειδή δεν άκουσα τον κύριο Τσασκόφσκι, ε, ελπίζω να μην τον επακαλύψω, να πω πάντως ότι ήταν μεγάλη ευχαρίστηση η συνεργασία μαζί του και την προηγούμενη εβδομάδα στη Βέρνη που είχαμε πολλές επαφές με Ελβετούς βουλευτές αλλά και με τον Ελβετό Πρόεδρο. Και νομίζω ότι καταλάβαμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους κανόνες της εταιρικής αγοράς και τη σχέση με το ελβετικό σύστημα. Να καταλάβουμε δηλαδή και ποιες είναι οι αρμοδιότητες καντονιών και ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτό πάντως που ήταν επίσης ενδιαφέρον είναι ότι τα καντόνια ενδιαφέρονται να αυξήσουν τη συνεργασία. Και στην επίσκεψη στη... συνειδητοποιήσαμε ότι ορισμένες ε, τοπικές ε, αυτοδιοκήσεις, έχουν ε, την δυνατότητα να αναλαμβάνουν ορισμένες πρωτοβουλίες, έχουν ορισμένες αρμοδιότητες επί της εσωτερικής αγοράς. Κάτι που συζήτησε με τους Ελβετούς ε, συναδέλφους και για το οποίο έλαβα μία σαφή απάντηση, αν και όχι επιθετική, ήταν ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες εισέγει μέτρα τα οποία δημιουργούν διακρίσεις κατά των υπηρεσιών από τρίτες χώρες. Εγώ είπα ότι ίσως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ακόμη και μεταξύ διαφορετικών καντονιών στην Ελβετία θα δημιουργούνταν προβλήματα εξαιτίας της διαφορετικής νομοθεσίας και ότι ίσως θα έπρεπε η Ελβετία να εξετάσει το θέμα και εσωτερικά. Γιατί ίσως τότε να διαπίστωναν ότι αν έλυναν τα εσωτερικά προβλήματα θα λύνονταν και αρκετά από τα προβλήματά τους με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Επίσης, άλλο θέμα. Το μοναδικό σημείο επαφής με την Ελβετία. Είναι κάτι που επίσης μας ενδιαφέρει στις συναλλαγές μας και ίσως να κάνω και μια σχετική τροπολογία για να επιστήσω την προσοχή σε αυτά τα θέματα γιατί νομίζω ότι όταν το αναφέραμε η αντίδραση ήταν θετική. Συμφωνεί σε αυτό και ο εισηγητής. Οπότε θα μπορούσαμε να γράψουμε κάτι πολύ γενικά βέβαια. Πάντως είδαμε ενδείξεις ότι τους ενδιαφέρει η διαδικασία, αλλά όχι οι επίσημες δεσμεύσεις, οι νομοθετικές δεσμεύσεις. Κάποια άλλα θέματα για τις χώρες ΕΟΧΑ και ΕΣΕΣ όσον αφορά την παροχή πληροφοριών εκ των προτέρων. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Όμως συμφωνώ με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι ότι η πρωτοβουλία που αποφασίσαμε να λάβουμε ως Επιτροπή ήδη ήταν πολύ σημαντική και διεύρυνε τα κανάλια επικοινωνίας μαζί τους. Θεωρώ ότι οι βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτές τις ε, επιτροπές ενημερώθηκαν αρκετά για τις δραστηριότητές μας και έτσι θα μπορούν να συνεισφέρουν με ιδέες τους και να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς εντός του ΕΟΧ που είναι ο βασικός μας στόχος. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπορ. Η κυρία Τέιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα είμαι σύντομη ε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τη γραμματεία για όλα αυτά που παρουσίασαν ε, με την έκθεση αυτή. Όταν έγινε λόγος για τη δημοκρατία και την άμεση δημοκρατία, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να εξηγηθεί το πώς ακριβώς ε, μέσα στο σύστημά μας υπάρχουν δυνατότητες να αντιμετωπιστούν κάποιες προκλήσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί υπάρχει και η αντιπροσωπεία με την Ελβετία, την Ορβηγία, την Ισλανδία και Ο συνάδελφος που ηγείται αυτής της αντιπροσωπείας βρίσκεται στη δική σας την ομάδα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε εξετάσει το θέμα όχι ως αντιπροσωπεία αλλά ως ε, ομάδα και αυτό θεωρώ ότι έτσι κάπως πρέπει να συνεχιστεί. Ο Ραφαέλ έχει μια πολύ καλή ισορροπία στην έκθεσή του. Αυτό πρέπει να τον αγνωρίσουμε και σίγουρα αυτό που πρέπει να προβάλλουμε είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε κήρυγμα στους Ελβετούς αλλά να αναζητήσουμε τρόπους ε, συνεργασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να συμφωνήσουμε και μετά να προχωρήσουμε γιατί δεν θέλω αυτή η έκθεση να ψηφιστεί εδώ και μετά να ξεχαστεί. Αυτό είναι κάτι που πάντα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ε, να θέλουμε την τελική πρόοδο θέλω ε, με αυτούς ε, που συναντηθήκαμε την περισμένη εβδομάδα να συνεχίσουμε την επαφή, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο μέλλον. Θέλω ε, να ευχαριστήσω όλους τους αρμόδιους και για την επισκέψη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελβετία. Επόμενη είναι η κυρία Βάιλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να κάνω πιο δύσκολη τη ζωή των συναδέφων από ότι είναι ήδη δύσκολη, αλλά εξεπλάγει για τα όσα ανέφερε ο κύριος Κρόιτσμαν, ότι υπάρχουν λέει εμπόδια λόγω της άμεσης δημοκρατίας στην Ελβετία, ώστε νομοθετήματα να εφαρμόζονται, νόμοι να υλοποιούνται. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουν σχετικά μικρό βαθμό άμεσης δημοκρατίας όμως καμιά φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο και θυμάμαι όταν είχαμε διαβουλευτεί και ήμουνα σε μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή όταν διαβουλευόμαστε για την ελευθερία κυκλοφορίας των εργαζομένων από τις κεντροανατολικοευρωπαϊκές χώρες και με ευχάριστο τρόπο εξεπλάγει ότι η, Ελβετή, η Ελβετία ήταν πολύ πιο γενναιόδορη και ρύθμισε αυτά τα πράγματα ταχύτερα και με πιο γενναιόδορο τρόπο από ότι η Γερμανία ή η Αυστρία που μέχρι σήμερα δεν έχουμε φτάσει εκεί και η Ελβετή χρόνια πιο πριν ε, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και άνοιξαν τα σύνορά τους. Ακόμα και αν κάποιες, κάποιοι περιορισμοί είναι ακόμα δυνατόν να εφαρμόζονται εκεί. Εξεπλάγει λοιπόν. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά, αν γίνεται, να ακούσω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δεν γίνεται σήμερα, ίσως στην τελική συζήτηση που θα διαξαχθεί την επόμενη φορά. Πώς δηλαδή αυτά τα εμπόδια βρίσκονται σε συσχετισμό με το θέμα της άμεσης δημοκρατίας και των ενώσεων και συλλόγων κτλ. Διότι υπάρχει ελπίδα ότι κάποτε στο εγγύς μέλλον η Ελβετία θα γίνει κανονικό τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα ήταν, αυτό θα ήταν ένα εμπόδιο όσον αφορά το συνταγματικό αυτό, τη συνταγματική δομή της ε, Ελβετίας. Δεν είναι κακή, κακές προθέσεις ή μη κακές προθέσεις, αλλά έχει σοβαρές επιπτώσεις σε αυτό το θέμα ίσως. Ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή επιπτωσεις αυτο το θεμα ισως από την νομική πλευρά να μας αποσαφηνίσει το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you. I guess we will have the possibility. Θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα εστερότερα να το κάνουμε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να προετοιμάσει μια τέτοια απάντηση για αυτή την ερώτηση. Επόμενο αγορητής, ο κύριο Σουάμπ. Παρακαλώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω φυσικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Για μένα και νομίζω και για κάποιους άλλους συναδέλφους είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι και προσωπικά μας αφορά. Και έγινε λόγος για την αντιπροσωπεία και για την Ελβετία όπου ε, είμαστε και συνάδελφοι μέλη. το θέμα αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε ασκηθεί, θα έλεγα. Έχουμε μια επικοδομητική έκθεση και συμφωνώ ότι στη σωστή, στα σωστά σημεία επελέγει η σωστή διατύπωση. Έχω μια ερώτηση προς τον εισηγητή σε σχέση με, τα, με την Ελβετία. Από ό,τι γνωρίζω δεν συμβαίνει ότι αυτό στο σημείο 7 η Ελβετοί είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την οδηγία περί παροχής υπηρεσιών. Από τη συμφωνία πλαίσιο του παρελθόντος ε, στο παρελθόν παραμένει και έτσι δεν υλοποιείται σε σχέση με την Ελβετία. Στο σημείο 13 το έχουμε και πάλι άλλη μια φορά. Αν αυτό θα μπορούσε να ρυθμιστεί ότι τα μέσα για την υλοποίηση από πλευρά Ελβετία μπορούν να προβλεφθούν, ακόμα και αν δεν είναι αυτό υποχρεωτική, δεν είναι δέσμευση, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, θα ήταν θετικό. Για το 10 δεν ξέρω αν είναι μεταφραστικό λάθο ή αν ίσω από την επιλογή των όρων και τη διατύπωση μπορεί να γίνει λίγο πιο σαφέ. Γράφει ο εισηγητή σωστά ότι διατυπώνει λέει ότι αυτά τα μέτρα κτλ. κτλ ιδιαίτερα αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να παρακολύονται στην Ελβετία. Το θα μπορούσαν είναι υπερβολικά επιφυλακτικό. Είναι σαφώς μια επιβάρυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμποδίζονται, ε, επιβαρύνονται. Αυτή η διατύπωση είναι υπερβολικά επιφυλακτική. Και ενδιαφέρον είναι φυσικά ότι αυτά τα θεσμικά θέματα με την Ελβετία αναφέρονται. Πρώτον στο σημείο 5. Στο σημείο 5 σε σχέση με το Κοινοβούλιο της ε, Ελβετίας να διαμορφώνει αυτά τα θέματα. Όμως κανονικά αυτό από τα κοινοβούλια των κρατών μελών επιφυλάσσει το δικαίωμα. Και αυτές οι μεικτές ε, αντιπροσωπείες είναι ε, σώματα, είναι όργανα τα οποία συζητούν ε, και κλεισμένων των θυρών και θα ήθελα να είναι δυνατό ένα πιο ανοιχτό πλαίσιο για αυτές τις αντιπροσωπείες ε, να μπορούν οι πληροφορίες ε, να δίνονται αυτές που στο Συμβούλιο και κλεισμένων των θυρών εξετάζονται και ποτέ δεν μας τίθενται στη δική μας διάθεση και αυτό θα ήταν κάτι σημαντικό. Κατά τα άλλα είναι εξαιρετική έκθεση και ευχαριστώ γι' αυτό. Thank Ευχαριστώ κυρία Γκέμπχαρτ. Η κυρία Γκέμπχαρτ ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ βρίσκω την έκθεση ισορροπημένη και καλή και μια καλή βάση για τη δουλειά μας εδώ. Θα ήθελα να, αναφέρω στο, να αναφερθώ στο σημείο 5 καταρχήν που το θεωρώ σημαντικό και σωστό διότι ακριβώς για τα κράτη ΕΖΕΣ και τώρα κάνω λόγο λιγότερο για την Ελβετία αλλά για τις υπόλοιπες χώρες ΕΖΕΣ. Διότι στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουμε εδώ πρέπει να εφαρμόζονται. Και γι' αυτό το βρίσκω σωστό και θεμητό και δίκαιο έγκαιρα τα νομικά κείμενα να είναι στη διάθεσή μας για να μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας και εμείς και έγκαιρα να ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται να εφαρμοστεί. Είναι κάτι το θετικό και πρέπει να το προωθήσουμε αυτό ως πρακτική. Και ξέρω από τους συναδέλφους σε σχέση με την Ορβηγία που είχαν συνέρθει και το συζήτησαν ότι και για αυτούς είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Και θα έλεγα ότι είναι κάτι το πολύ θετικό και ωραίο. Θα ήθελα να θέσω μια επερώτηση για το σημείο 16 και εδώ υπομειδιώντας θα ήθελα να αναφέρω για το τελευταίο τμήμα χαιρετίζει την πιο πρόσφατη προσαρμογή της, της ελβετικής ε, νομοθεσίας όσον αφορά το θέμα Κασίτε Νομίζω αυτό το ξέρουμε απ' έξω πια, το έχουμε διαβάσει τόσες φορές. Όμως ακριβώς εξίσου συχνά έχουμε ακούσει και διαφορετικές ερμηνείες για αυτή την υπόθεση, για την ομολογία δηλαδή του δικαστηρίου για το Cassis de Dijon. Και πρέπει να στραφώ στον εισηγητή και να ρωτήσω ποια από αυτές τις ερμηνείες είναι εκείνη που εννοεί εκείνος και έχει υπόψη. Διότι αυτό αφήνεται ασαφήνιστο, δεν έχει αποσαφινιστεί. Και έτσι θα ήθελα να ξέρω τι βρίσκεται πίσω από αυτή τη διατύπωση ουσιαστικά από αυτό το εδάφιο. Διότι πολλές συζητήσει γίνονται και πάρα πολλά πράγματα ερμηνεύονται και εντάσσονται σε αυτή την ομολογία, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, χωρίς να είναι όμως αυτά όλα βάσιμα. Θέλω να μου πείτε περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Ευχαριστώ. Okay, Ευχαριστώ και τώρα μπορούμε να ακούσουμε την Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο, αλλά και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Στο παρελθόν η Κομισιόν έχει εκφράσει την εκτίμησή της για την έκθεση αυτή και έχουμε αναφέρει αρκετές φορές ε, την άποψή μας. Θεωρούμε ότι η έκθεση αναφέρεται σε πολλές θετικές και αρνητικές πτυχές των τομεακών ε, συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελβετία και σωστά υπογραμμίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Όπως ε, ήδη έχει αναφερθεί, αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει είναι την, ενιόμορφη, την ομοιόμορφη εφαρμογή. Και εδώ μιλάμε για στατικές συμφωνίες που δεν λαμβάνουν υπόψη τους το νέο κεκτημένο. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί έτσι οι Ελβετοί φορείς Ορισμένες φορές απολαμβάνουν περισσότερα προνόμια από ότι οι Ευρωπαίοι φορείς. Κάτι που θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιο για τους Ευρωπαίους. Δεν έχουν υπάρξει αλλαγές από το 2008. Δεν έχει ολοκληρωθεί καμία νέα συμφωνία με την Ελβετία για την πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όπως θυμάστε, το 2008 είχαμε συμπεράσματα της Συμβουλίου που ζητούσαν ότι οποιοδήποτε νέα μελλοντική συμφωνία με την Ελβετία θα έπρεπε να λάβει υπόψη της αυτά τα στοιχεία. Άρα εμείς θα λάβουμε υπόψη μας τις συστάσεις της έκθεσής σας και κυρία Στήλερ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα ξεχάσουμε την έκθεση, δεν θα την καταχωνιάσουμε στα ντουλάπια γιατί έρχεται σε μία πολύ καλή χρονική συγκυρία. Το Συμβούλιο πρόκειται να αναθεωρήσει τα συμπεράσματα του 2008 για τις σχέσεις με τις χώρες ΕΖΕΣ ε, το δεύτερο εξάμεινο του έτους και επίσης όπως ε, γνωρίζετε, παρόμοιες ε, συζητήσεις όπως αυτές που γίνονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται και στην Ελβετία. Για παράδειγμα, εντός του μηνός θα υπάρξει μία έκθεση της ε, Συνομοσπονδίας, ενώ επίσης περιμένουμε εντός του θέρους και ε, την έκθεση Μακβάλτερ. Άρα, νομίζω ότι θα φανούν σαφώς οι παράμετροι που ισχύουν και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μελλοντικά βήματα. Βεβαίως, οι ελβετικές αρχές είναι αυτές που θα αποφασίσουν τι μορφή θα ήθελαν να έχουν οι σχέσεις μας. Μία ακόμη πτυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω και που αναφέρθηκε από ομιλητή αφορά τη συμμετοχή της Ελβετίας στην ε, διαμόρφωση των αποφάσεων. Να σας υπενθυμίσω ότι γίνεται αυτό στην Νορβηγία επειδή υπάρχει αυτόματη έγκριση του κεκτημένου. Άρα είναι λογικό να ισχύει αυτό για την Νορβηγία όπως και για την Ισλανδία και το Λίχτενστάιν εφόσον αυτομάτως πρόκειται να υιοθετήσουν αυτό το κεκτημένο. Η διαφορά με την Ελβετία είναι ότι η Ελβετία έχει μόνο στατικές συμφωνίες, δεν εγκρίνει αυτομάτως το κεκτημένο, άρα το θέμα αυτό είναι πιο πολύπλοκο. Μια άλλη ερώτηση. Ομολογώ ότι χρειάζεται περισσότερη προετοιμασία για να μπορέσω να την απαντήσω. Αφορά το θέμα της δημοκρατίας και της εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε με την Ελβετία για να βρούμε τρόπους για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Αν και θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην ε, συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Απλά πρέπει να γνωρίζουμε τις συνέπειες των αποφάσεων. Αυτή τη στιγμή ισχύουν κάπου συμφωνίες όπου υπάρχει ρήτρα γκυλοτίνας. Δηλαδή, αν καταψηφιστεί σε ένα δημοψήφισμα μια συμφωνία, σταματάει η ισχύς όλων των υπολείπων συμφωνιών. Βεβαίως αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε με τις ελβετικές αρχές, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε μαζί και με τα υπόλοιπα θέματα που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Ολοκληρώνω εδώ και επαναλαμβάνω πολύ ενδιαφέρουσες οι υποδείξεις της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε και μία ερώτηση για την αρχή του Κασίντε Τζιζιόν. Ευτυχώς ε, δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω εγώ αυτή την απόφαση Κασίντε Τζιζιόν γιατί αυτό το έπραξε ήδη πριν από μένα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. γιατί αυτό ε, μπήκε σε σχετισμό με το Reinheitsgebot ε, την αρχή περικαθαρότητας και ούτω καθεξής. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα ελβετικά δικαστήρια δεν είναι αναγκασμένα να δεχθούν αυτή την απόφαση και αυτό πραγματικά είναι σχεδόν ανήκουστο. Γιατί, γιατί υπάρχει αυτή η περίεργη σχέση μεταξύ ημών κατόπιν τούτου οι Ελβετοί ε, δεν δέχονται κάποια στοιχεία νομοθεσίας ε, δικά μας. Η ερμηνεία δική τους μπορεί να είναι διαφορετική και δεν δεσμεύονται από την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό λοιπόν μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα γιατί δεν υπάρχει ε, αποδεκτή ερμηνεία και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχει νομική ασφάλεια ως εκ τούτου. Όλο και περισσότερο ελβετικά δικαστήρια στις αποφάσεις τους παραπέμπουν ε, στις ερμηνείες που δίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα ελβετικά δικαστήρια οποτεδήποτε αποφαίνονται ε, κάνουν αναφορά ε, στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και αυτό είναι καλό. Σε πάρα πολλές λοιπόν περιπτώσεις έχουν ε, αναφέρει, έχουν κάνει επίκληση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κυρίως για την περίπτωση Κασίς de Τα ελβετικά δικαστήρια συμφωνούν με αυτή την απόφαση, αλλά εμεί θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα χέρια, γιατί το όλο θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια των Ελβετών δικαστών και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει ενιαία εφαρμογή. Πάντω, στην πραγματικότητα, η ενιαία εφαρμογή, η εφαρμογή και στις δύο πλευρές, ε, υφίσταται, γιατί σας είπα, οι δικαστές είναι ανοιχτοί. Τώρα, όσον αφορά την ενημέρωση, κοιτάξτε, η συνθήκη της Λιζαφώνας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ε, δίνει τη δυνατότητα τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να ενημερώνονται περισσότερο. Και εμείς αυτό το εφαρμόζουμε πρακτικά. Δηλαδή, καλούμε τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων για να έχουν συζητήσεις με μας. Και κάτι άλλο εφόσον υπάρχουν στενές σχέσεις ε, με την Ελβετία και τις χώρες ΕΟΧ, θα πρέπει να τους ενημερώνουμε, να ενημερώνουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια το συντομότερο δυνατόν. Γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ομοθεσία. Όσον αφορά τώρα την διαμόρφωση των αποφάσεων, ε, είναι σημαντικό να καλούμε τους αδέλφους να αποφαίνονται. Αυτό έγινε με τους Νορβηγούς, καλό θα ήταν να γίνει και με τους Ελβετούς. Να τους καλέσουμε εδώ, σε αυτήν την Επιτροπή, ε, στη συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και ξέρετε πολύ καλά, μετά τη Λισαβόνα αλλά και πριν από αυτήν υπήρχε η συναπόφαση. Άρα δηλαδή η διαμόρφωση υποφάσεων λαμβάνει χώρα και εδώ. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να ανοίξουμε λίγο περισσότερο τις ε, πόρτες μας. Στο σημείο υπερθμών 10 και σε αυτά που είπε ο Ανδρέας, ε, πράγματι ε, διπλωματική θέλουμε να είναι η διατύπωσή μας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών. Ίσως πρέπει να αλλάξω εδώ λιγάκι το ύφος, δεν έχω πρόβλημα, θα το δω. Τώρα, όσον αφορά σε αυτά τα ειδικά σχόλια, αυτά είχα να πω και περιμένουμε βέβαια τις ε, τροπολογίες ε, με τους ε, σκιώδεις συγητές. Θα δουλέψουμε πάνω στις συμβαστικές προτάσεις και όπως σας είπα και εγώ θα αλλάξω μόνος μου κάνα δύο πράγματα γιατί γι' αυτό έκανα το σχέδιο πριν από δύο μήνες μετά είχαμε την ακρόαση, κάναμε το ταξίδι, διαβουλεύσεις θα το αλλάξω λοιπόν σε κάποιο βαθμό το σχέδιό μου αλλά όχι ριζικά κόκκινη γραμμή είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι πρέπει να καταδείξουμε το δρόμο του μέλλοντος και τουλάχιστον να καλέσουμε και τις δύο πλευρές να ε, διερευνήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Όπως σας είπα πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά είναι η 7η Ιουνίου και ε, μέχρι τότε λοιπόν ε, θα συνεργαστώ με τους σκιώδης και θα λάβουμε υπόψη μας τις τροπολογίες που εντωμεταξύ θα έχουν κατατεθεί, θα τις λάβουμε υπόψη μας όσο πιο σοβαρά μπορούμε. Ευχαριστώ όλους για αυτή την εξαιρετική συζήτηση. Αναγγέλλω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 7η Ιουνίου στι 18.06 το απόγευμα. Και τώρα πρέπει να ολοκληρώσουμε το δημόσιο τμήμα, ανοιχτό τμήμα αυτής της συνεδρίασης. Θα συνεχίσουν οι συντονιστές σας. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.